Σας καλωσορίζω, καλωσορίζω το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτολή, Επιτροπή και θα δώσω τον λόγο στα δύο αυτά όργανα σε λίγο. Έχουμε την κοινή συζήτηση για τους μηχανισμούς ενίσχυμένης οικονομικής διακυβέρνησης. Έχουμε μια δήλωση του Συμβούλιο διότι θα μας μιλήσει για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής της 7ης Μαΐου 2010. Θα έχουμε επίσης προφορικές ερωτήσεις στο Συμβούλιο και την Επιτροπή για την Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 στο πλαίσιο της σημερινής χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και για τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στη στρατηγική ΕΕ 2020 και τη διακυβέρνησή της και προφορικές ερωτήσεις στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή για τη σημασία της στρατηγικής ΕΕ 2020 στο πλαίσιο της σημερινής χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Ο πρώτος ομιλήτης εξ ονόματος του Συμβουλίου δίνω τον λόγο στον ε, κύριο Καριντά, υφυπουργό. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όλοι γνωρίζουμε ότι διανύουμε μία περίοδο ε, εξαιρετικών και ε, οικονομικών αναταραχών. Πριν από λίγους μήνες ε, ξεκίνησε αυτό